και της ευκολότερης πρόσβασης στη χρηματοδότηση και στους όρους πλαίσιο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε, Υπουργέ. Και έτσι φτάνουμε στο πέρας της συζήτησης σε αυτού του σημείου. Έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ και θα περάσουμε στο επόμενο σημείο στον Οργανισμό Ανάπτυξη και Συνεργασία στην Ευρώπη. Ενίσχυση του ΟΑΣΕ και ο ρόλος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο, ο πρώτος ομιλητής εξ ονόματος της ε, Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και της είπα της ε, εκπροσώπου Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, ο Πρόεδρος Τσαστέλ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ε, με ιδιαίτερη τιμή ε, ε, θα εκφωνήσω την ομιλία με εξονόματος τη κυρίας Άστον ενώπιόν σας. Ε, ξέρετε ότι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των 56 κρατών μελών του ΟΑΣΕ θα μεταβούν στο Άστανο για τη Σύνοδο Κορυφής και 35 χρόνια μετά την πράξη του Ελσίνκη, 25 χρόνια μετά το χάρτη του, Παρι, του Παρισιού, και 11 χρόνια μετά τη δήλωσή της Κωνσταντινούπολης ε, βλέπουμε πόσο σημαντική είναι αυτή η σύνοδος γιατί χρειάζεται μια νέα όθηση. Ε, ο ΑΣΕ ορισμένοι αμφισβήτησαν τη χρησιμότητά του. Ε, κάποιοι θεώρησαν ότι δεν ήταν σε θέση να καθαρίσει τα ερήπια του ε, ε χρού πολέμου και κάποιοι ε, θεωρούν ότι δεν είναι αποτελεσματικός οργανισμός. Το 2008 ο πρόεδρος Μετβέτεφ απέφθινε έκκληση να αναθεώρηση της αρχιτεκτονικής της ασφάλειας στην Ευρώπη και έτσι ε, επανατροφοδοτήθηκε ο διάλογος ε, για τον ΟΑΣΕ και άρχισε η διαδικασία της Κέρκυρας. Ε, ο ΟΑΣΕ, χωρίς να αποκλείουμε και άλλα ενδεδειγμένα φόρα τέτοιων συζητήσεων, έχει πάντως ανακτήσει την εμπιστοσύνη όλων και παίζει κρίσιμο ρόλο και εξάλλου η πρόταση του κυρίου Ρουσέκ το επιβεβαίωσε αυτό. Η διάσκεψη αναθεώρησης ε, μας ε, επέτρεψε να οριοθετήσουμε τη διαδικασία. Στη Βιέννη τώρα ε, έχει τεθεί υποδιαπραγμάτευση το τελικό κείμενο που θα υποβληθεί στη συνέχεια στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. Έχει τρία μέρη αυτό το έγγραφο. Πρώτον αρχές, ε, κανόνες και δεσμεύσεις του ΑΣΕ. Δεύτερον, κοινέ προκλήσεις και προτεραιότητες. Και τέλος, ένα κομμάτι πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό που αφορά τη δράση του ε, θα πρέπει να είναι βανάγνωστο δε αυτό το έγγραφο για όλους τους πολίτες ε, της Ευρώπης ε, ε, και έχουμε ιδιαίτερε φιλοδοξίε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω και άλλα μέλη του ΑΣΕ. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μία ε, κοινή κοινότητα, δηλαδή θα έχουμε την ευρασιατική κοινότητα, ενιαία κοινότητα, χωρί καμία διαχωριστική γραμμή, όπου θα ζουν όλοι οι πολίτε σε ασφάλεια, όπου θα επιλύονται ειρηνικά ε, οι συγκρούσει και οι αρχέ και οι κανόνε που είναι το κεκτήμενο του ΑΣΕ θα γίνονται σεβαστέ. Αυτό πρέπει να στόχος της Συνόδου θα προκύψει και μία έντολη και ένας οδικός χάρτης από αυτή τη Σύνοδο. Ένα σχέδιο δράσης. Ε, η ασφάλεια χαρακτηρίζει τον ΟΑΣΕ και αυτές οι τρεις διαστάσεις θα πρέπει να συνυπολογιστούν και να βρεθεί μία ισορροπία μέσα σε αυτό το έγγραφο προκύψει από τη Σύνοδο. Τονίζεται αυτό μέσα στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου και οι Υπουργοί Εξωτερικών ε, όταν ε, συναντήθηκαν τον Ιούνιο Ιούνιο ε, τόνισαν ότι υπάρχουν πολύ σημαντικέ πηγέ μεταξύ των οποίων πολιτικο-στρατιωτική. Ο εξυγχρονισμό του εγγράφου τη Βιέννη ε, για τα μέτρα ασφαλεία ε, και εμπιστοσύνη αποτελούν ενθαρρυντικό στοιχείο. Τώρα για τη συνθήκη για τι συμβατικέ δυνάμει στην Ευρώπη είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητά του, Συνεχίζονται έντονε οι διαπραγματεύσει και αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων είναι εκείνοι που θα πρέπει να δώσουν την απαραίτητη όθηση για να προχωρήσουμε δυνατότητα του ΟΑΣΕ να ανταποκριθεί σε αυτές τις τρεις προκλήσεις θα πρέπει να ενισχυθεί ούτω ώστε να έχουμε έγκυρη ε, προειδοποίηση, επίλυση των συγκρούσεων, ανοικοδόμηση, Έχουμε τις προτάσεις όλων των εταίρων και η δημιουργία μιας τέτοιας κοινότητα ε, τι σημαίνει ότι θα πρέπει να δούμε στη στο, ε, στο στην Ουκρανία θα πρέπει ε, να δούμε τα ερήπια αυτών των συγκρούσεων, πώς μπορούμε να τα καθαρίσουμε και κυρίως να εκφράσουμε μια κοινή βούληση, πολιτική βούληση για να επιληθούν αυτές οι συγκρούσεις και για να ε, δείξουμε... Ε, όταν ε, λύσουμε τις παρελθούσες συγκρούσεις ότι μπορούμε στο μέλλον να αντιμετωπίσουμε τις νέες διασυνοριακές συγκρούσεις σε συνεργασία με άλλους ε, συναρμόδιους ε, διεθνείς φορείς. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιμένει το ενεργειακό θέμα να εξεταστεί υπό το πρίσμα της επίλυσης των ε, συγκρούσεων. Επίσης, η οικονομική του πρέπει να ενισχυθεί, οι αρχές για την καλύτερη διακυβέρνηση ε, να πληρούνται, το θέμα της ασφάλειας για την ε, ενεργειακή τροφοδοσία θα πρέπει επίσης να πληρούνται. Έχουμε ένα ε, κοινό έδρανο αξιών ε, επί του οποίου θα οικοδομήσουμε και αυτήν τη νέα κοινότητα ασφαλείας και χρειαζόμαστε ε, νέα μέσα για να προχωρήσουμε. Θα, υπο... Ε, θα συμπεριληφθούν στο έγγραφο που θα υποβληθεί στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων και κατόπιν θα προκύψουν συστάσεις του ΟΑΣΕ ε, τη... για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ΑΣΕ είναι ένα απαραίτητο βοήθημα για όλα τα κράτη-μέλη και επίσης επιμένει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη σημασία της ελευθεροτυπίας και των ελευθέρων εκλογών στη ζώνη του ΟΑΣΕ. Επίσης, το Γραφείο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Δημοκρατίας θα πρέπει να έχει ένα ενισχυμένο ρόλο και να διατηρηθεί η αυτονομία του επίσης ε, οφείλουμε να ενισχύσουμε τη δράση της ΕΙΠΑ του εκπροσώπου κυρίως στον τομέα της ελευθερίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ Υπουργέ Σαστέλ και τώρα θα δώσω το λόγο στους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων. Ε, πρώτα απ' όλα, εξ του ΕΛΚ, ο κύριος Γκζίμπ ε, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ είπα κύριε Πρόεδρε. Ακούσαμε από τον εκπρόσωπο της υψηλής εκπροσώπου για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και έχουμε επίσης και το ψήφισμα το οποίο συνέταξε ο Λίμπο Ρότσεκ, ο Ευρωβουλευτής Λίμπο Ρότσεκ, που λέει ότι η διαδικασία της Κέρκυρας χρειάζεται μια νέα όθηση. Αυτό είναι κάτι το οποίο και η ίδια η ύπατη εκπρόσωπος έχει διαδηλώσει. Ο ΟΑΣΕ θα μπορούσε να είναι ένας πραγματικά πάρα πολύ σημαντικός οργανισμός για την επίλυση περιφερειακών συγκρούσεων για τα προβλήματα των εθνοτικών μειονότητων και τη δημοκρατικοποίηση στα κράτη-μέλη του. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την ισορροπία μεταξύ του πολιτικο-στρατιωτικού πυλώνα, του περιβαλλοντικού πυλώνα και του ανθρώπινου πυλώνα η παραδοσιακή έννοια της σκληρής στρατιωτικής δύναμης ως βάση για την ασφάλεια είναι πολύ σημαντική, αλλά είναι σημαντική και η οικονομική, η κοινωνική ασφάλεια και η ασφάλεια εφοδιασμού σε τρόφιμα. Ο ΑΣΕ θα πρέπει να πράξει περισσότερο στον τομέα αυτό. Να παίξει μεγαλύτερο ρόλο στην παρακολούθηση των εκλογών με παρατηρητές και το το πρόγραμμα για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα επίσης έχει ε, παίξει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στις χώρες μέλη του ΟΑΣΕ. Είναι μια δραστηριότητα η οποία αξίζει υποστήριξης, αλλά όλα αυτά τα οποία πράττει ο ΟΑΣΕ δεν μπορούν <clears throat> να περιοριστούν στην απλή διαμεσολάβηση. Ο ΟΑΣΕ είναι ένας φορέας ο οποίος επιτρέπει στις χώρες να λάμπουν δια της προεδρίας τους. Παραδείγματος χάρη, ο ρόλος του Καζακστάν στην τωρινή κρίση που έπληξε το Κυργιστάν και η διαμεσολάβησή του μεταξύ του Ορκμενιστάν και Ουσμπεκιστάν ήταν πάρα πολύ χρήσιμη. Η, διάσκεψη κορυφής του Δεκεμβρίου στην Αλμάτι θα πρέπει να βοηθήσει να μπορέσουμε να εγκρίνουμε τον μελλοντικό χάρτη του ΟΑΣΕ. Και γι' αυτό θέλω να υποστηρίξω το ψήφισμα το οποίο έχει διατυπώσει ο κ. Ρούτσεκ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει και ο πρόεδρος. Αντιπρόεδρε κ. Λίμπορ Ρούτσεκ, έχετε τώρα το λόγο. Για τρία λεπτά, κύριε Αντιπρόεδρε. Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. Φέτος γιορτάζουμε τον 35η επέτειο από την τελική πράξη του Ελσίνκη. Η διαδικασία του Ελσίνκη συνεισέφερε στην ιστορική αλλαγή που σημειώθηκε στην Ευρώπη η οποία κάποτε χωριζόταν από την εποχή του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου από τον ψυχρό πόλεμο. Τώρα που συμβιωθηκε στην ευρωπη η οποια καποτε χωριζοταν απο την εποχη του δευτερου παγκοσμιου πολεμου απο τον ψυχρο πολεμο τωρα που εληξε πια ο χωρισμός αυτός από το σιδηρούν παραπέτασμα πρέπει να δούμε αν έχουν επιτευχθεί όλοι οι στόχοι της διαδικασίας του Ελσίνκη. Ακόμη σημειώνονται εθνικές, εθνοτικές διαμάχες μεταξύ γειτονικών χωρών και δεν έχουν ριζώσει όλες οι δημοκρατικές αξίες σε όλες τις χώρες υπάρχουν και προκλήσεις ασφαλείας όπως η τρομοκρατία, το δουλεμπόριο η παράνομη διακίνηση ναρκωτικών. 35 χρόνια λοιπόν μετά το Ελσίνκι και 11 χρόνια μετά από τη διάσκεψη της Κωνσταντίνου Πόλεως πρέπει εδώ στην Ευρώπη να υπάρξει μία αναθέρμανση, μία αναζωογόνηση, μία μεταρρύθμιση. Η διαδικασία της Κερκύρας έδειξε σε ποια κατεύθυνση πρέπει να κινηθούμε και το ίδιο πρέπει να πράξει και η επόμενη επικείμενη διάσκεψη του Δεκεμβρίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει κάνει ορισμένες συστάσεις, προτάσεις για τη διάσκεψη αυτή να συζητήσει και να εγκρίνει ένα σχέδιο δράσης για την πρόληψη των σειράξεων, για τη διαχείριση των κρίσεων και για την ανοικοδόμηση μετά από τέτοιες εκρήξεις. Έτσι θα μπορέσουμε να δείξουμε το, να ανοίξουμε το δρόμο για να δημιουργηθεί μια χάρτα, οδικός χάρτης για την ασφάλεια. Ο ΟΑΣΕ, όπως είπαν και άλλοι, είναι αναπόσπαστο τμήμα της ευρωατλαντικής και ευρωασιατικής δομής ασφαλείας. Πρόκειται για κράτη που πάνε από το Βανκούβερ μέχρι το Βλαδιβοστόκ. Και η οικονομική, στρατιωτική, περιβαλλοντολογική, νομική συνεργασία μεταξύ των όλων αυτών των χωρών πρέπει να διασφαλιστεί. Η Ευρώπη, ενδυναμωμένη πια από τη συνθήκη της Λισαβόνας, πρέπει να βοηθήσει να συνεισφέρει σε αυτού του είδους τη συνεργασία γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα εξ ονόματος των φιλελευθέρων, όχι των σοσιαλιστών. όχι, το ακούσαμε με σοσιαλιστε. σοσιαλιστές. Των φιλελευθέρων, των φιλελευθέρων, για δύο λεπτά, η κυρία Ανιέλη Γιάτενμάκη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο ΟΑΣΕ ανέκαθεν ήταν πολύ σημαντικός οργανισμός ε, που έχει ε, του σεβασμού όλων και τώρα τον, σήμερα τον χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ. Συχνά αυτός ο οργανισμός μας επιτρέπει να έχουμε πρόσβαση σε ζώνες κρίσης, ενώ άλλοι οργανισμοί αντίστοιχοι δεν έχουν τέτοια πρόσβαση. Χρειαζόμαστε λοιπόν τον ΟΑΣΕ, τον χρειαζόμαστε στην Κεντρική Ασία. Χρειαζόμαστε την υποστήριξή του για αστυνομικές επιχειρήσεις, για την καταπολέμηση του εμπορίου ναρκωτικών, ναι, για την κατοχήρωση των συνόρων Επίσης είναι μοναδική και η ανθρωπιστική του δραστηριότητα. Σε αυτό το καλάδι, σε αυτό το κομμάτι του ΟΑΣΕ, στην ανθρωπιστική δράση, έχουμε δει νέους τρόπους καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων και επίσης ε, βλέπουμε, παρατηρήσαμε ενίσχυση των δυνατοτήτων ε, αδύναμων κρατών. Πάντως, οι δράσεις εστιάζονται στις αστυνομικές επιχειρήσεις με τη χρήση παραστρατιωτικών ε, δυνάμεων. Ενεργοδραστηριοποιείται ο ΑΣΕ σε διάφορους τομείς ε, που σχετίζονται με την ασφάλεια και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να ε, ακολουθήσει το παράδειγμα του ΟΑΣΕ στις ε, δικές της επιχειρήσεις γιατί πρώτος φτάνει συχνά ο ΟΑΣΕ, είναι και πιο πεπειραμένος οργανισμός, έχει πεπειραμένους ε, εμπειρογνώμονες Η ισχύ του ΟΑΣΕ βέβαια εξαρτάται από τη βούληση των κρατών μελών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να εκτιμήσουμε το έργο του ΟΑΣΕ. Ευχαριστούμε για τους πρασίνους, ο κύριος Μπιτκόφερ. Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος ε, Σαστέλ. Ο κύριος Σαστέλ μίλησε για μια νέα δυναμική του ΟΑΣΕ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ήθελε να συμβάλλει στο να εξευρεθεί αυτή η νέα δυναμική. Το ψήφισμα το οποίο έχουμε ενώπιον μας σήμερα υπό την ηγεσία του παντιπρόεδρου κ. Ρούτσεκ και το οποίο υποστηρίζεται από μια ευρύτατη πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει μια πολύ προοδευτική αντιμετώπιση για το ρόλο του ΟΑΣΕ στο μέλλον. Χρειάζεται μια νέα όθηση. Αυτό έχει λεχθεί από πάρα πολλούς ότι είναι απαραίτητο να μπορέσει να προωθηθεί ο οασέ σε πολλούς τομείς. Έχουμε την ε, ε, κρίση του Αμερικανικού Αντιπροέδρου για το ρόλο του ΟΑΣΕ που τον θεώρησε ιδιαίτερα θετικό, αλλά χρειαζόμαστε επιπλέον και μια καλύτερη στοχοθεσία για την διαδικασία που θα οδηγήσει στην χάρτα του ΟΑΣΕ. Και οι τρεις διαστάσεις του ΟΑΣΕ πρέπει να ενισχυθούν και ιδιαίτερα το Γραφείο για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Θέλουμε όμως να προχωρήσουμε και σε νέα εγχειρήματα. Παραδείγματο χάρη, υπάρχει το ερώτημα του κατά πόσο θα είναι δυνατό στο μέλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, στα πλαίσια της ΚΕΠΑ, της ε, κίνησης της πολιτικής εξωτερικών θεμάτων και ασφάλειας, να αναλαμβάνει αποστολές με εντολή του ΟΑΣΕ. Στην περίπτωση της παραδείγματο χάρη, θα ήταν πάρα πολύ θετικό να υπήρχε μια τέτοια δυνατότητα και να μπορούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να συμμετάσχει σε ενέργειες μαζί με τους Ρώσου. Εξάλλου, <clears throat> όπως αναφέρθηκε προηγουμένως από τον Αντιπρόεδρο Ρούσεκ, πρέπει να δώσουμε και συγκεκριμένου στόχους στη διαδικασία της Κέρκυρας που οδηγεί στην εκπόνηση μια συνολικής χάρτας στα πλαίσια του ΟΗΣΕ για τα θέματα ασφάλειας. Νομίζω ότι είναι μια σωστή απάντηση στις προτάσεις της ρωσικής πλευρά, η οποία ήθελε να προωθήσει μια νέα συζήτηση για την ασφάλεια στον διατλαντικό χώρο. Για μένα ο ΑΣΕ θα παραμείνει απαραίτητος για να εξασφαλιστεί η αρχιτεκτονική ασφαλείας στον ευρωπαϊκό και ατλαντικό χώρο και ελπίζω ότι η διαδικασία που ακολουθείτε θα είναι και αυτή η επιτυχία. Σε ευχαριστώ πολύ ο κύριος Τένοκ για τους συντηρητικούς. Ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, ο ΑΣΕ παίζει ένα σημαντικό και ολοένα αυξανόμενο ρόλο για να προωθήσει την ειρήνη και τη σταθερότητα στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Το γεγονός ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε, η Ρωσία και χώρε Κεντρική Ασία είναι πλήρη μέλη του ΩΣΑ, αυτό αυξάνει την αξιοπιστία και το εύρο του φορού, φορέα αυτού. Από το Βανκούβερ μέχρι το Βλαδιβοστόκ λειτουργεί ο ΑΣΕ. <clears throat> Ξεπερνάει πια το Συμβούλιο της Ευρώπης ως ο κυριότερος χώρος για τη συζήτηση της δημοκρατίας και φυσικά παίζει και σημαντικό ρόλο για την παρακολούθηση εκλογών. Για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την κατάσταση του κράτους δικαίου παίζαν σημαντικό ρόλο. Σε χώρε όπω η Γεωργία και η Μολδαβία, οι αποστολέ του ΟΑΣΕ βοήθησαν πάρα πολύ στο να σταθεροποιηθούν οι κοινωνίε αυτέ, οι οποίε είχαν τραυματιστεί από παγωμένε σειράξει και πρόσφατε αντιπαραθέσει Το Καζακστάν που έχει την Προεδρία του ΟΑΣΕ έχει ανυψώσει το προφίλ του φορέα αυτό και έχει εστιάσει την προσοχή μα στην Κεντρική Ασία, ιδιαίτερα στο θέμα τη ασφάλεια και του αγώνα κατά τη διεθνή τρομοκρατία. Χωρί αμφιβολία υπάρχουν πολλέ δυνατότητε για να αναπτύξουμε τι σχέσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση περαιτέρω μαζί με τον ΟΑΣΑ. Αλλά όταν σφυριλατούμε αυτή την εταιρική σχέση, πιστεύω ότι η ύπατη εκπρόσωπο θα πρέπει να κάνει τι απαραίτητε προσπάθειε να μην υπάρξει επικάλυψη προσπαθειών και σπατάλη χρημάτων φορολογουμένων σε μια εποχή λιτότητας και θα πρέπει να συντονιστεί καλύτερα ο ΑΣΕ με την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα την ΚΕΠΑ και το ΝΑΤΟ για την εταιρική σχέση για την ειρήνη. Και τέλο, θα ήθελα να προτείνω οι δύο φορεί, το Συμβούλιο τη Ευρώπη και ο ΑΣΕ, θα μπορούσαν να σκεφτούν να συγχωνευτούν και έτσι θα γλιτώσουμε πάρα πολλά λεφτά. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να σα υπενθυμίσω ότι πρέπει να παραμείνετε μέσα στον χρόνο ομίλησής σα, γιατί τα μεσάρικτα θα φύγουν οι διερμηνείς. Και δεν θέλω να μιλάμε μέχρι τι 2 η ώρα στα αγγλικά. Ο κύριο Σόλτ για την ΚΟΕ 2 λεπτά. Η πολιτική μου ομάδα, λέει ο κ. Σόλτ, χαιρετίζει το γεγονό ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά από πάρα πολύ καιρό έχει αντιμετωπίσει και πάλι το θέμα του ΟΑΣΕ και επομένω τι ε, σχέσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση με τον ΟΑΣΕ, τη διαδικασία του Ελσίνκη και την ανάπτυξη μηχανισμών για τι σημερινέ προκλήσει. Ότι όλα αυτά μπορούν να τύχουν θετική απάντηση. Η έκθεση του κ. Ρότσερ τονίζει <clears throat> ότι δεν μπορούν οι, Ευρώπη και οι να είναι αντίπαλοι, αλλά θα πρέπει να λειτουργούν από κοινού και θα πρέπει να αναλάβουν τις απαραίτητες αρμοδιότητες. Για μένα, με, με τη διάσκεψη της Αστάνα, υπάρχουν μερικά στοιχεία τα οποία θέλω να υπογραμμίσω. Χρειαζόμαστε μια κοινή στάση στην Ευρώπη για την πολιτική στρατηγική του μέλλοντος και για την ε, Ήπειρο της ε, Ασίας, η οποία σήμερα αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα ασφαλείας. Θα πρέπει να έχουμε μια διαρθρωμένη συζήτηση για τα θέματα αυτά, η οποία θα, διαμορφω... θα πρέπει να διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο από τα κρατημένα, ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συγκεκριμένε αποφάσει για τον τομέα τη ασφάλεια και του αφοπλισμού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ΚΕΠΑ στον τομέα αυτό θα πρέπει να αντιμετωπίσουν παράλληλα και το θέμα τη ασφάλεια εφοδιασμού σε ενέργεια και τη κλιματική αλλαγή, ώστε να μπορούμε να έχουμε πραγματικά διαρθρωμένη συνεργασία στου τομεί αυτού. Ακολουθεί κυρία Δύο λεπτά. Πρόεδρε, Υπουργέ Σαστέλ, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα στην παρέμβασή μου να επιμείνω στο κεντρικό ρόλο των αποστολών παρατήρηση εκλογών για την ενίσχυση και των σχέσεων μας με τον ΟΑΣΕ, αλλά και γενικότερα για την ενίσχυση τη εξωτερική μας δράση για να υπάρχει σεβασμός των ατομικών πολιτικών δικαιωμάτων που είναι αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να κατοχυρώσουμε την ακαιρεότητα των εκλογικών διαδικασιών. Αυτό έχει ζωτική σημασία για την εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ένωσης. Από, με αυτές τις αποστολές ε, παρατήρηση εκλογών λοιπόν θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε, είναι προς συμφέρον μας, με τον ΟΑΣΕ. Η υπηρεσία εξωτερικής δράσης ε, νομίζω απαιτεί διαδικασία στενής συνεργασίας ανάμεσα ε, στο Γραφείο Δημοκρατίας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ και τον, του αντίστοιχου τμήματο της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. Έτσι δεν θα έχουμε επικάλυψη και θα ενισχύσουμε την εξωτερική δράση της Ένωσης στη ζώνη του ΟΑΣΕ. Αυτή η συνεργασία θα, θα πρέπει να γίνεται πριν κατά τη διάρκεια και μετά την αποστολή ε, για να προετοιμαστεί καλά η, ε, αποστολή για να υλοποιηθεί σωστά και να υπάρξει και παρακολούθηση μετά. Ε, επίσης ε, θέλω να τονίσω το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εκπροσωπούμε ε, τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε αιρετοί εκπρόσωποι, οπότε πρέπει εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εκμεταλλευτούμε αυτό το ατούπο έχουμε να παρακολουθούμε ε, τις εκλογές ε, τρίτων χωρών. Επίσης αναγνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι η οικονομική και η περιβαλλοντική δράση του ΟΑΣΕ γιατί ε, αυτά επηρεάζουν συχνά και τη σταθερότητα και την ασφάλεια. Την πραγματογνωμοσύνη του ΟΑΣΕ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να την εκμεταλλευτούμε και επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα οικονομικά και περιβαλλοντικά στοιχεία που ε, θα ε, εξασφαλίσοντας έτσι το αίσιο πέρας ε, των αποστολών μας. Ενισχύοντας τη συνεργασία λοιπόν με τον ΟΑΣΕ και χάρη στην παρουσία των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου νομίζω ήδη έχουμε ενισχύσει την ναι. εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπακούντας στα όσα επιτάσσει η συνθήκη της Λισαβόνας. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Νταπάλζη. Σας ευχαριστώ. Θέλω να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία. Διότι όλοι γνωρίζουμε ότι μέσα στην Ευρώπη εκτός από την Ένωση το Συμβούλιο της Ευρώπης και ο ΑΣΕ είναι οι σημαντικότερες οργανώσεις που έχουν διαθέτουν τεράστια εμπειρία για τη διαχείριση διεθνών ή εθνοτικών σειράξεων και διαφορών. Και έτσι μπορούμε να δούμε ποια είναι ακριβώς η προστιθέμενη αξία, η σημασία του ΟΑΣΕ σας ανέφερα ήδη για τις διαφορές και σειράξεις. Το γεγονός ότι ο ΑΣΕ έχει έναν ύπατο αρμοστή, ο οποίος συχνά παρεμβαίνει και δρά διαμεσολαβητή σε τέτοιες σειράξεις, είναι κάτι που διευκολύνει πολύ, που προωθεί μάλλον την ασφάλεια των μειονοτήτων το 90% των σειράξεων που σημειώνονται είναι εθνοτικές. Πρέπει λοιπόν να εμπνευτούμε και εμείς στην Ένωση από την εμπειρία του ΟΑΣΕ. Για τους Ρωμά ας πούμε, ε, ο ΟΑΣΕ υπήρξε πρωτοπόρος σε πολλά προγράμματα και θα ήθελα να τονίσω τα προγράμματα αυτά. Όταν προετοιμάζουμε εμείς τη στρατηγική μας για τους τσιγκάνους πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας την εμπειρία του ΟΑΣΕ. Υπάρχει η δήλωση της Κοπεχάγης του 1990 για την, το δικαίωμα μειονοτήτων σε αυτοδιάθεση. Επίσης, όταν ακούμε τους εκπροσώπους του, τον εκπρόσωπο του ΑΣΕ που είναι υπεύθυνο για την ελευθεροτυπία, βλέπουμε ότι μιλάει πιο ελεύθερα για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων και άλλων δικαιωμάτων μέσα στα κράτη-μέλη από ότι εμείς οι ίδιοι και γι' αυτό υποστηρίζω τόσο πολύ τη συνεργασία μας με τον ΟΑΣΕ. Ευχαριστούμε η κυρία Χαουτάλα. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Θα ήθελα να, στηρί... να υποστηρίξω αυτά που είπε ο συνάδελφος Μπουτικόφερ για την εξισορρόπηση των τριών διαστάσεων που διαθέτει ο ΑΣΕ. Πρέπει την ανθρώπινη από αυτές τις διαστάσεις να τονίσουμε ιδιαίτερα. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί η έκθεσή μας λαμβάνει υπόψη της και το γεγονός ότι η χώρα της τωρινής προεδρίας το Καζαχστάν πρέπει να σεβαστεί και εκείνη τις βασικές αρχές του ΑΣΕ, εν ώψη της διάσκεψης του που επίκειται. Δεν είναι ικανοποιητικά τα πράγματα. Εκεί υπάρχουν πολλές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κλπ. Uh, ε, επίσης σημειώνω ότι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δέχονται πολλοί συνάδελφοι ότι πρέπει να παίξει πιο ενεργό ρόλο. Η κοινωνία των πολιτών είναι πολύ θετικό ότι μπορεί και πρέπει να συμμετέχει στην ε, διοργάνωση της διάσκεψης του Αστάν, της Αστάν. Ευχαριστούμε πολύ. Μιγκάλ, ο κύριος Μιγκάλσκι. Για ένα λεπτό. Χαίρομαι που χρησιμοποιείτε τα πολωνικά κύριε Πρόεδρε. Εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εμείς οι Πολωνοί και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι θα πρέπει να προωθήσουμε το ρόλο της, του ΟΑΣΕ, ιδίως όταν τα συμφέροντά μας συμπίπτουν με αυτά του ΟΑΣΕ. Παραγωγός χάρη στην Γεωργία, η υπερπληστερία, στο σχέδιο έξι σημείων του Σαρκοζή για την Γεωργία κτλ. Δίκιο έχει η κυρία Χάουταλα, το ίδιο ισχύει και για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά πάνω από όλα θα πρέπει να θυμόμαστε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας φορέας και η σχέση μας με τον ΟΑΣΕ δεν θα πρέπει να μας κάνει να βασιζόμαστε στον ΟΑΣΕ για τη λήψη αποφάσεών μας. Είναι ευρύτατη η συμμετοχή στον ΟΑΣΕ, δεν είναι μοναχα η Ευρωπαϊκή Ένωση που συμμετέχει εκεί. Και η, η συνδέση με τον ΟΑΣΕ μπορεί να είναι αντιπαραγωγική σε μερικές περιπτώσεις. Ακολουθεί ο κύριος Σόγκορτ. Ευχαριστώ. Από την ίδρυσή του, ο ΑΣΕ θεωρούσε ότι το πρωταρχικό του καθήκον ήταν η έγκυρη προειδοποίηση και πρόληψη ε, των συγκρούσεων. Ε, έχουμε ένα γραφείο για τις εθνικές μειονότητες μέσα στον ΟΑΣΕ, ώστε να αποφεύγονται οι εντάσεις ανάμεσα στην ε, πλειοψηφία και την μειοψηφία. Δηλαδή έγκαιρη διπλωματική προειδοποίηση, έτσι ονομάζεται αυτό. Νομίζω ότι τα όργανα του ΟΑΣΕ μπορούν να παίξουν ζωτικό ρόλο. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ε, η πράξη για την επίσημη γλώσσα στη Σλοβενία όταν αποπειράθηκε, είπα ότι εκπρόσωπος να διαμεσολαβήσει, δεν υπήρξε καμία εξέλιξη. Δεν τελεσφόρησε αυτή η προσπάθεια και αυτό συνεχίζει να αποτελεί πηγή εντάσεων γιατί συνιστά διακριτική μεταχείριση και παραβιάζει διάφορες ε, διεθνείς ε, συμφωνίες όπως έχει ήδη συμπεράνει η Επιτροπή της Βιέννης. Ίσως να προσεγγίζαμε Now Ας περάσουμε στο ΚΑΤΣΙΑΗ, ο κύριος Χίγκιν. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μας μιλάνε για τον ΟΑΣΕ λέγοντας ότι ε, προβάλλουμε την ελευθερία και τα πολιτικά δικαιώματα. Υπουργείο Σαστέλ, ωραία. Πώς το ε, συνδυάζεται αυτό με το ότι το Καζακστάν έχει αναλάβει την Προεδρία φέτος και ε, στην πρωτεύουσα την Αστάνα θα γίνει σύνοδος το Δεκέμβριο. Γνωρίζετε ότι τα πολιτικά δικαιώματα ε, το, στο Καζακστάν παραβιάζει. δεν υπάρχει η ελευθερία των ε, μέσων μαζικής ενημέρωσης, οι ακτιβιστές σαπίζουν στις φυλακές και το Σεπτέμβριο ήμασταν στην αποστολή στο, όπου διαπιστώσαμε βάναυση μεταχείριση των κρατουμένων. Πριν από δύο εβδομάδες ο πρόεδρος Μπαρόσα τι κάνει. Ε, βγάζει το κόκκινο χαλί για τον πρόεδρο Ναζερμπαϊγέφ για τον υπεύθυνο όλων αυτών, χωρίς κανένα επικριτικό σχόλιο. Γιατί ε, οι συμφωνίες για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο κανονίζουν τι θα γίνει στη Σύνοδο, στην Αστάνα. Πρέπει να είμαστε σοβαροί και να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Αν το εννοείτε ότι θέλετε να ε, υπερασπιστείτε τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα των πολιτών του Καζακστάν ευχαριστούμε. Ο κύριος θέλει για να απαντήσει εξ ονόματος της κυρίας Άστον. Ευχαριστώ. κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς που παρεδέρωσαν για την ποιότητα του διαλόγου και θα διαβιβάσω στην Λέδη Άστον τις προτάσεις σας, ιδίως ό,τι αφορά την ορθολογικοποίηση των ε, μέσων και την καλύτερη χρήση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και σε ό,τι αφορά τα θέματα συνεργασίας μας. Εξάλλου, <clears throat> δεν νομίζω ότι χρειάζεται να επανέλθω σε αυτά τα οποία ανέφερα στην αρχή της παρέμβασής μου, γιατί πολλοί βουλευτές ανέφεραν πράγματα ταυτόσιμα από αυτά που είπα. Για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Καζακστάν. Έχετε δίκιο να υπογραμμίσετε αυτή την ε, πτυχή. Πολύ το πράξατε απόψε. Πολύ σημαντικά είναι όλα αυτά για την Ευρωπαϊκή Ένωση υπενθυμίζουμε αυτό το πρόβλημα σε όλες τις επαφές μας με τους ηγέτες του Καζακστάν. Την ανάγκη να συνεχιστούν οι προσπάθειες σε ό,τι αφορά την αναβάθμιση των πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και της δημοκρατικοποίησης. Το θέμα της δημοκρατίας αναφέρθηκε από ότι, αντίθετα από ό,τι φαίνεται να λένε ορισμένοι στην τελευταία ε, επίσκεψη του κυρίου Ναζαρμπάιεφ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να κλείσω λέγον ότι η διάσκεψη της Αστανά με την ηγεσία του Καζαχστάν θα μας δώσει μια μεγάλη ευκαιρία να ξεπεράσουμε τα προβλήματα του παρελθόντος, να αναπτύξουμε μια κοινότητα ασφάλειας από το Βανκούβερ ως το Βλαντιβοστόκ, όπως είπατε προηγουμένως, και να αποδηθούμε σε νέες αποστολές που θα μας οδηγήσει σε ένα περιβάλλον ασφάλειας που αρμόζει στον 21ο αιώνα. Χαιρόμαστε που το Κοινοβούλιο υποστηρίζει την πρωτοβουλία αυτή τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειαζόμαστε αυτή την εκπεφρασμένη υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να αναβαθμίσουμε την αξιοπρέπεια του ατόμου, τι ελεύθερε εκλογέ και την εξασφάλιση της ενέργειας σε διεθνικών απειλών καθώς και την αρμονική συνεργασία σε ένα αηφόρο περιβάλλον. Ελπίζουμε ότι με τον τρόπο αυτό θα περάσουμε σε μια νέα φάση της γόνιμης ιστορίας του ΟΑΣΕ, ιδίω στην Αστάνα και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αναλάβει και θα υπομειστεί τις ευθύνες της. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Συνάδελφοι, λίγη εδώ αυτή η συζήτηση. Θα ψηφίσουμε αύριο. Τώρα το επόμενο θέμα.